Chers collègues, euh, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σα. Ευχαριστώ όλους όσους μπόρεσαν να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί που ξεκινάνε οι εργασίες μας. Είμαστε στο σημείο 15. Τον λόγο θα τον ε, δώσω στην ε, Νάντια Χίρσ για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της ε, που αφορά την αντιμετώπιση της πρόορης αποχώρησης από το σχολείο. Είναι μια γνωμοδότηση την οποία συντάσσουμε για την Επιτροπή Πολιτισμού. Νάντια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. zuerst einmal... Ε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή μου. Innerhalb der EU 2020. Στη στρατηγική 2020 περιλαμβάνεται αυτή και ορίζεται και ως στόχος η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου να παραμείνει, ε, να πέσει στο κάτω του 10%. Σε πολλά κρατημέλη έχουμε ποσοστά πολύ περισσότερα, πολλές φορές πάνω από 20%. Και θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα στοχευμένα και με βάση τη δημογραφική αλλαγή. Να παροτρύνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας. Οπότε, ε, στόχος μας θα πρέπει να είναι και αυτή η ομάδα, όχι μόνο ο δικός μας και των κρατών μελών. Είναι μια ομάδα μαθητών που έχει μεγάλο δυναμικό και δεν θα πρέπει να καταλείπει ορίσει στο σχολείο. Δεν υπάρχει κανένας νέος που να μην έχει καμία ικανότητα, κανένα προσόν, καμία δεξιότητα. Μπορεί κάποιο να είναι καλύτερο σε κάτι άλλο και να μην προσφέρεται το σχολικό σύστημα για να αναδείξει ε, την αξία του, τι ικανότητε, τα προσόντα του. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, είναι ιδιαίτερη ομάδα που αξίζει την προσοχή μα και στη στρατηγική 2020, όπω είπα προηγουμένω. Για τον λόγο αυτό, όπως και στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας είπα, ο στόχος είναι το 10% και παρακάτω. για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε καλούς εργαζομένους, για να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε σωστά. Αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη και στα εθνικά τους μεταρρυθμιστικά προγράμματα έχουν ε, προτείνει ορισμένα μέτρα. Τι γίνεται λοιπόν στα κράτη-μέλη. Γιατί καλό είναι να έχουμε στρατηγική ε, και στόχους ε, στο 2020, αλλά ε, καλούνται τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Ähm, είναι πολύ βασικό λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο τρόπος εκμάθησης και διδασκαλία στο σχολείο, να ξαναδούμε δεχομένως τον κλασικό τρόπο λειτουργίας και παροχής γνώσης στο σχολείο Και επίσης και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μετακπαιδεύονται. Και η εκπαίδευση στις παιδαγωγικές ακαδημίες, στα πανεπιστήμια ε, να γνωρίζουν ε, πώς ε, θα αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση, πώς θα τη μεταδίδουν καλύτερα στους μαθητές, όχι το κλασικό μάθημα παράδοση από καθέδρας. και καταλαβαίνουμε ότι είναι σε θέση οι μαθητές εκείνοι, είναι εκείνοι που καταλήγουν το σχολείο χωρίς ε, δίπλωμα, χωρίς ε, τίτλους. Και όταν το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας ήδη ε, κάπως χαμηλότερο, αυτό είναι ένας παράγον που επιδεινώνει την κατάσταση. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν καν την ευκαιρία, τη δυνατότητα ακόμα και το ήθελα να τελειώνουν το σχολείο. Παράδειγμα, Πολύ συχνά το έχουμε ξαναδεί και στη στρατηγική για τους Ρωμά ή ε, σε παιδιά που οι δεν έχουν επίσημα έγγραφα ε, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει και εκεί να τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ένα δίπλωμα, ένα πολιτήριο σχολείου, αλλιώ δεν θα έχουν ποτέ τη δυνατότητα να ορίζουν το μέλλον τους. Αυτά. Ε, χρειάζεται λοιπόν αλλαγή και στην οτροπία του σχολείου, αλλά και των θεσμών. Μεγαλύτερη ευελιξία. Με προσοχή να κοιτάξουμε αυτό το θέμα, πώς θα αξιοποιήσουμε ε, τους μαθητές αυτούς. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο μεταξύ και μάλιστα συνδυασμένο, όχι μόνο για εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αλλά γενικά για όλους τους νέους, για να μπορούν να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Μία ομάδα λοιπόν από αυτό το σύνολο των νέων είναι οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Και ε, τα διαρθωτικά ταμεία μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και το κοινωνικό ταμείο, επί παραδείγματι, για να φτάσουμε και στο στόχο της ε, στρατηγικής 2020. Θα πρέπει στοχευμένα να διοχετεύουμε και πόρους εκεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτά εισαγωγικά και σύντομα για την γραμμοδότηση. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού, όπω είπατε, και η δυσκολία ποια είναι. Στι 8 Ιουνίου θα πρέπει να ψηφίσουμε εμεί τι δικέ μα τροπολογίε, αλλά ήδη στι 9 του μηνό ψηφίζεται η έκθεση στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ λίγο αυτό το διάστημα, μία μέρα μόνο, για να μπορέσουμε να διαβιβάσουμε τι ιδέε μα στην Επιτροπή Απασχόληση. Από την Επιτροπή απασχόληση δηλαδή στην Επιτροπή Πολιτισμού. Καλό λοιπόν να φροντίσουμε νωρίς να ε, βρούμε συμβαστικές τοπολογίες για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε για την Επιτροπή Πολιτισμού. Με χαρά θα συνεργαστώ με τους και ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκουτιέρες έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ. Σύντομα, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπε η συγκήτρια, την οποία και ευχαριστώ για τη εργασία της στην έκθεση αυτή. Ε, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μερικές ιδέες που θεωρώ σημαντικές. Συμφωνούμε όλοι ότι η εκπαίδευση, η μόρφωση είναι η βάση για την ισότητα των ευκαιριών. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος κανείς ε, είναι, όσο περισσότερο έχει μορφωθεί στο σχολείο, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει να βρει δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, και θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε πώς αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις συγκεκριμένες χώρες, ε, θα το λύσουμε γιατί είναι μάστιγα πραγματικά. Πρέπει να στείλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ότι έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην παιδεία οι πολίτες. Δεν θα πρέπει να το απεμπολούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισότητα των ευκαιριών να είναι κανείς καλά ε, προετοιμασμένος η έλλειψη μόρφωσης είναι μειονέκτημα, είναι επιβαρυντικός παράγων ε, και οδηγεί περισσότερο προς τη φτώχεια. Στην έκθεση αυτή αναφέρουμε τρεις ιδέες. Ε, και πρόληψη και επέμβαση και ε, αντιμετώπιση, αντιστάθμιση αν θέλετε. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μειωθούν οι δείκτες πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Τώρα στα πλαίσια των αρμοδιότητων της δική μας Επιτροπής θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στο σχολείο. Μας λένε όλοι ότι χρειάζεται ένα νέο σχολείο ε, προσαρμοσμένο στη νέα κοινωνία που να ποντάρει ε, στην κοινωνική ενσωμάτωση ε, και στη συμβίωση. Όλοι μας λένε ότι ε, όταν έχουν προβλήματα τα σχολεία ένταξης, συμβίωσης κάποιων πολιτών, είναι μεγαλύτερη η πρόορη εγκατάλειψη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα στοιχείο για το σχολείο. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε την ιδέα, και είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή, να συμφιλιώνεται ο επαγγελματικός βίος με το σχολικό και το ε, εργασιακό. Δηλαδή όταν σε μια οικογένεια υπάρχουν προβλήματα ε, συνδυασμού της εργασίας των γονέων με τον οικογενειακό βίο υπάρχουν προβλήματα και στα παιδιά και πρόορη εγκατάλειψη. Κάτι άλλο που προσάπτω εγώ στη γνωμοδότηση αυτή είναι το θέμα της αποζημίωσης ή της αντιστάθμισης. Έχω κάποιες αμφιβολίες εδώ. Δηλαδή κάποιοι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, καλό είναι να τους βοηθούμε να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, αλλά δεν μπορούμε να φτιάχνουμε προγράμματα και να τους στέλνουμε μηνύματα ότι μπορεί να είναι αυτή η οριστική λύση, η εναλλακτική λύση. Δηλαδή φύγει από το σχολείο και θα βρει δουλειά από τα κοινοτικά προγράμματα, θα τους βοηθήσουμε. Όχι. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι είναι δική του υποχρέωση να συνεχίσουν το σχολείο, να τελειώσουν το σχολείο. Και εμείς δεν θα πρέπει να φτιάχνουμε μπαλώματα για να μπαλώνουμε κάποια κακή κατάσταση, αλλά να τη διορθώσουμε. Γιατί τους στέλνουμε σε επισφαλείς μορφές εργασίας και τελικά στη φτώχεια. Καλύτερα λοιπόν να μορφώνονται και όχι να εγκαταλείπουν το σχολείο και εμεί να ερχόμαστε να τους σώζουμε βρίσκοντας δουλειά σε εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει τις του, τους, πούμε, τη σχολική του εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν τα μεικτά προγράμματα που επιτρέπουν να εντάσσονται μεν στην αγορά εργασία, αλλά να συνεχίζουν το σχολείο είναι τα καλύτερα. Γιατί έτσι ε, θα βρουν καλύτερη δουλειά, θα έχουν πιο πολλά προσόντα και πιο ε, ποιοτική απασχόληση και όχι αυτές τις εμβαλωματικές λύσεις που προτείνουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριος Μπάχ και μετά κύριος Μάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως Επιτροπή νομίζω έχουμε δύο δυσκολίες. Επικουρικότητα, δηλαδή αρμοδιότητα των κρατών μελών το ένα και το δεύτερο ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το έγγραφο εργασίας και την πρόταση για σύσταση στο Συμβούλιο νομίζω είναι σε καλό δρόμο Καλή είναι η προσέγγιση, ε, ψάχνει τους λόγους ε, γιατί ε, εγκαταλείπουν πρόωρε μαθητές στο σχολείο, αναλύει την κατάσταση στα κράτη-μέλη, γιατί δεν είναι πάντα ίδια. Και... κοιτάει πώς μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν προγράμματα και στρατηγικές για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Τώρα να και στα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά τους για να δούμε πώς θα ανταποκριθούν. Η Ισπανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία απέχουν πάρα πολύ ε, από ε, τα benchmark από τη, τα ορόσημα αν θέλετε, που έχουμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε να εργαστούμε και στη στρατηγική του 2020 γι' αυτό. Κατά τα άλλα έχουμε δύο προβλήματα αυτοί οι μαθητές που φεύγουν πρόωρα από το σχολείο λείπουν και από την αγορά εργασία γιατί δεν έχουν τα προσόντα, δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν καταρτιστεί όπως θα έπρεπε και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε εργαζομένους από χώρε εκτός της Ένωσης. Και ε, είναι και μεγάλο το οικονομικό τίμημα. Και επιπλέον έχει και κοινωνικές επιπτώσεις αυτό μακροπρόθεσμα. Είναι σύντομη η γνωμοδότηση της κυρίας Χέρς, την καλωσορίζω και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί της. Νομίζω ότι ως Κοινωνική Επιτροπή θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς συνδέεται το σχολείο με την αγορά εργασίας, αλλά και να προωθήσουμε την ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα. Επίσης, να κοιτάξουμε αυτό το ζήτημα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν καλά παραδείγματα που μπορούμε να τα ακολουθήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε και στην έκθεση. Και κάτι άλλο ε, είναι η ατζέντα για νέα προσόντα και δεξιότητες και το πρόγραμμα νεολαία σε δράση. Και στη στρατηγική του 2020. Ε, επαναλαμβάνω να την εντάξουμε γιατί είναι απολύτω απαραίτητη για την ευρωπαϊκή αγορά εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τόμασμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Άτια Χέρι. Έχει κάνει πολύ καλή έκθεση και πάρα πολύ επικεντρωμένη στα ουσιώδη. Εντάξει, η, ε, η παιδεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει φροντίσει να δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ε, μαθητές να βγουν από αυτή την κατάσταση, να μην εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται σχολείο και επάγγελμα, σουπ, που στα γερμανικά είναι και ως λογοπαίγνιο και δίνει τη, λέξη όθηση. Τους δίνουμε λοιπόν την όθηση να μπορέσουν να συνδυάσουν το σχολείο και το επάγγελμα. Ε, και βλέπουμε το ιστορικό της οικογένειας. Πολλές φορές ε, το επίπεδο της οικογένειας, ε, το μορφωτικό είναι πολύ χαμηλό και πολλές φορές, για να μην πω ε, πάντα, ο μόνος που ξυπνούσε το πρωί και σηκωνόταν ήταν ο μαθητής για να πάει στο σχολείο από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους, να τους δώσουμε τα εφόδια, να τους δώσουμε τα προσόντα και μια αυτοπεποίθηση που δεν παίρνουν από την οικογένειά τους. Και να καταλάβουν ότι μπορούν να πάνε ένα πτυχίο, να τελειώσουν ένα σχολείο, να μορφωθούν και να τους πούμε ότι εσύ δεν είσαι απόκλειος της κοινωνίας από χέρι. Έχεις ευκαιρίες και αξιοποιείς έτσι. Εκεί βοηθάει το κοινωνικό ταμείο. Ε, στο σημείο 9 που αναφέρει στη στοχευμένη αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Αντί για διαρθρωτικά ταμεία δεν μπορούμε να πούμε ρητά ε, το κοινωνικό ταμείο και προτείνει το 8 και τη θέσπιση ενό πρότυπου σχεδίου. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια. Καλά κάνει και το προτείνει, αλλά δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτά που ήδη ισχύουν στα κράτη-μέλη ή σε ένα κράτο-μέλη. Που έτυχαν πολύ. Έτσι κι αλλιώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαστήρι και προσπαθούμε ε, με τις βέλτιστες πρακτικές να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν έχουμε ακόμα αναγνωρίσει όλη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη. Και τελευταίο, πολύ σωστά είπες ότι οι νέοι έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό ε, και δυνατότητες από ε, ό,τι ορισμένοι τους ε, αναγνωρίζουν. Και το πτυχίο, το, το δίπλωμα, το πολιτήριο σημαίνει κάτι. Πέρα από την κοινωνική αποκατάσταση είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, θέμα αξία. Ξέρω όλος ότι ε, μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του με εφόδια και ε, το βοηθάει πολύ. Αυτά, δύο-τρεις παρατηρήσεις και προτάσεις θα κάνω και εγώ με τροπολογίε, να είσαι βέβαια γι' αυτό. Ε, κυρία Τσουρινάν και μετά η κυρία Μωρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην όλη διαδικασία. Κατά πρώτον, να πω ότι το θέμα αυτό βρίσκω δύσκολο να προκαλέσει διαφωνίες στην Επιτροπή μας. Ξέρουμε ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα. Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να μορφώνονται και δεν διαφωνεί κανείς ότι το Στόχο αυτό θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή εμβέλεια εδώ, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να συμμετέσχουν τελικά στην αγορά εργασία και στην οικονομία γενικότερα. Αληθεύει, όπω υπόθηκε, ότι είναι ζήτημα που καλύπτεται την επικουρικότητα. Όμω αν το σκεφτείτε, Γι' αυτό έχει καλυφθεί και από τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Θα έχει τεράστιε συνέπειε για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Από κοινωνική πλευρά αλλά και από οικονομική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συζητηθεί και εδώ σήμερα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω ότι η καταπολέμηση της πρόορας εγκατάλειψης στο σχολείο υπήρξε ένας στόχος από χρόνια, ήδη από την στατική της Λισαβόνας, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Για να μην πω ότι έχουν αντιστραφεί οι όροι. Δηλαδή σε κάποιες χώρες τα ποσοστά για την πρόορη εγκατάλειψη έχουν ξεπεράσει το 30%, ενώ ο μέσος όρος για την, το 13% μάλλον το 30% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ο μέσο όρος έχει ξεπεράσει το 14%. Κάποια κάτι μέλη δεν εργάζονται αρκετά σκληρά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει επισημάνει στην σχετική τη έκθεση. Ε, παραθέτω εδώ, μόνο ορισμένα κράτη ακολουθούν συνεκτική και σφαιρική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν την πρώτη κατάληψη του σχολείου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τα κράτη-μέλη που μπορεί να έχουν μεν φορολογικέ δυσκολίε, αλλά αυτό ακριβώ δεν πρέπει να το Δημοσιονομικέ δυσκολίε αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούν το θέμα αυτό. Εδώ θέλουμε να συνεχιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως είπε και το Συμβούλιο χρειάζεται κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για αποτελεσματικές πολιτικές και για καλύτερη συμπερίληψη στα εθνικά προγράμματα βάσει της στρατηγικής του 2020. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις συνέπειες της πρόορας εγκατάλειψης του σχολείου, δηλαδή τι συμβαίνει αν αφήσουμε το πρόβλημα αυτό να διαιωνίζεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε σοβαρό κίνδυνο να αυξηθεί η φτώχεια και το να καταπολεμήσουμε την πρώην εγκατάλειψη πραγματικά είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων. Αυτό είναι ένα μέτρο καθοριστικής σημασίας, ώστε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια πολίτες να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να πετύχουμε έτσι ένα στόχο της στατική του 2020. Τέλος, θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των φίλων σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτό δεν αφορά βεβαίως ε, εδώ τόσο πολύ τις γυναίκες, όσο περισσότερο τα νεαρά αγόρια. Του νέου άντρε, διότι τα ποσοστά του είναι πιο αυξημένα τι στατιστικέ για την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και μπορεί να δημιουργήσουμε μια νέα τάξη νεαρών ανδρών με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και πολύ λίγε ευκαιρίε και δυνατότητε να συμμετάσχουν στην αγορά εργασία στο μέλλον. Είναι ένα σημαντικότατο λοιπόν πρόβλημα. Θα πρέπει να το έχουμε διαρκώ υπόψη. Σα ευχαριστώ για τη συζήτηση και ε, ανυπομονώ να συμμετάσχω στο όσο θα γίνουν τον επόμενο μήνα σχετικά. Ευχαριστούμε. Κυρία Μωρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ, όπως οι προηγούμενοι, και να συγχαρώ την εισηγήτριά μας. Εδώ ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημεία. Κατά πρώτον, σε σχέση με όσο είπε η κυρία Τουρούνεν, ε, συμφωνώ απολύτως ως προς το ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κάτι μέλη. Πίεση, λοιπόν, για να... γιατί βλέπουμε ότι δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν ε, οθούν τους νέους να φτάσουν στην υποχρεωτική ηλικία σχολικής εκπαίδευσης. Μπορούμε να συνεχίσω φαντάζομαι γιατί τα μικρόφωνα λειτουργούν. Οι νέοι λοιπόν με τη συνενοχή των ε, κρατών μελών αποκλείονται ουσιαστικά από το σχολείο. Άρα το σχολικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών μελών επιτρέπει στους νέους, τους δίνει ακριβώς την δυνατότητα να φεύγουν από το σχολείο πριν από την συμπλήρωση της υποχρεωτικής ηλικίας εκπαίδευσης. Μπορούν βεβαίως να φύγουν από το σχολείο χωρίς να πάρει τη μόρφωση, αλλά πριν την υποχρεωτική ηλικία είναι κάτι που το επιτρέπουν τα ίδια τα κάτι μέλη. Σε αυτή την περίπτωση ακριβώς δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω απολύτω και νομίζω ότι είμαι και πιο ε, μαχητική σε αυτό το σημείο από ότι η Εμιλή Εδώ υπάρχει πραγματικά ανεπάρκεια από την πλευρά των κρατών μελών ω προ τι υποχρεώσει του. Επίση υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη ισορροπία και ανισότητα μεταξύ κοριτσιών και αγοριών εδώ. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα θέματα ανακατηγορία ε, αγοριών και κοριτσιών ουσιαστικά διότι στα περισσότερα κράτη έχουμε την τάση να πετάμε από το σύστημα τα αγόρια από ό,τι τα κορίτσια. Διότι ακριβώ τα αγόρια δεν αντέχουν να πλήττουν στο σχολείο. Γίνονται ταραξίες ε, πιο εύκολα και, και έτσι τα κράτη πιο εύκολα εξωθούν εκτός του σχολείου τα αγόρια. Αυτό γιατί κάθονται πιο ήσυχα στην τάξη του σχολείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν δυσκολεύονται και εκείνε. διότι μπορεί και να μείνουν χωρί να μάθουν τίποτα. Και δεν σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν καλύτερα σε συστήματα επανένταξη, όπω έλεγε ο κ. Μαν. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μια σοβαρή, μια πραγματική μελέτη για όλα τα σημεία αυτά. Το τρίτο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια τάση μαζικοποίησης τη εκπαίδευση, Αλλά κάτι που δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και το δείχνουν αυτό οι στατικέ που περιέγραψε και ο κ. Μαν, είναι η εξατομίκευση. Όλοι οι νέοι ε, που έχουν δυσκολίε θα πρέπει να εποφεληθούν από στρατηγικές εξατομικεύσεις ακριβώς στα πλαίσια των ε, εκπαιδευτικών μας πολιτικών. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να εμείνουμε στην ε, έκθεσή μας. Τέλος, ε, μια τελευταία παρατήρηση. Έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία επιτρέπουν τους νέους να σχεδιάσουν προσωπικά προγράμματα κινητικότητας, επανένταξης, ώστε να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Ε, κάποιες φορές ακριβώς χάνουν την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, στην προσωπικότητά τους. Οπότε τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να γίνουν ένας πραγματικός μοχλός, ώστε οι νέοι, πέραν των γλωσσικών δυσκολιών ή προβλημάτων, να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Και με την ευρωπαϊκή κινητικότητα, με το άνοιγμα προς την Ευρώπη, να μπορέσουν να αυξήσουν τις δυνατότητες επανένταξης. Και όπως έλεγε και ο κύριος Μαν, στην εκλογική μου περιφέρεια έχω συζητήσει με νέους που δεν έχουν τα απαραίτητα μορφωτικά προσόντα, ζουν σε γειτονιές ε, δύσκολες, ε, μπορεί να είναι και σε κέντρα κοινωνικής ε, προστασίας, και του έχουν επισημάνει ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν έπειτα την επανένταξη σε επιχειρήσει και την ε, εργασιακή, τον επαγγελματικό βίο. Αυτό είναι ένα πραγματικό μοχλός, ε, ένα εργαλείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι συνάδελφοι που να ζητούν το λόγο. Έχει και πάλι το λόγο η συγγετρία κυρία Χίρ. Ευχαριστώ πολύ ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και για τις προτάσεις σας. Ε, εντάξει, με χαρά να δεχτώ τις προτάσεις για να βελτιώσω τα σημεία. Στο σημείο 3 προσπάθησα να πω ε, ότι θα πρέπει να μας αναφέρουν τι κάνουν τα κράτη-μέλη, αν κάνουν κάτι δεν έχω πρόβλημα να το διατυπώσω και με μεγαλύτερη σαφήνεια. Γιατί είναι και δική μας δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, θέτουμε καμιά φορά το δάκτυλο επί του τύπο των ύλων ε, για να επισημαίνουμε τα κακό κείμενα, αλλιώ δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ τη στρατηγική 2020. Και πολλέ φορέ εμεί τα ακούμε, ενώ αυτά είναι τα κράτη-μέλη που δεν ε, εφαρμόζουν αυτά που πρέπει. Κάτι άλλο, στο σημείο 6, η διάσταση του φύλου νομίζω είναι πραγματικά κομβική και θα πρέπει να το επεκτείνουμε ίσως. Εγώ ξέρετε έχω πρόβλημα όπως όλοι χαρακτήρων πρέπει να τηρήσω τη γνωμοδότηση σε κάποιο πλαίσιο. Μπορούμε να το αναφέρουμε με διαφορετικό τρόπο και να αναφέρουμε αγαπητέ Τόμας Μαν και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρω ότι στη δική μου περιφέρεια είναι ήδη πολλά τα καλά προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό που είναι κρίμα ε, είναι ότι έχουμε πολλές φορές ωραία προγράμματα που αποδίδουν, αλλά δεν τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν προβάλλονται σωστά. Ίσως είναι θέμα επικοινωνίας και διαφήμισης αυτό. Να ανταλλάσσουμε και καλές πρακτικές και εμπειρίες και προγράμματα. Λοιπόν, γενικά το θέμα δεν είναι επίμαχο, είναι μεγάλη η συμφωνία, αλλά και αυτή τη συμφωνία ε, που έχουμε να αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε επιτέλους και να φροντίσουμε το 2020 να έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον να φτάσουμε το στόχο μας έστω και με τρόπο στοιχειώδη. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, μην το κάνουμε και συνήθεια, αλλά Θέλω να είσαστε εφάνταστοι, χωρίς υπερβολές όμως. Διότι δεν έχουμε και βέβαια και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την ε, υποβολή των τροπολογιών ε, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να τις ε, εξετάσουμε τις τροπολογίες. Επομένως, καλό θα είναι να περιοριστείτε στα ουσιώδη. Προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών σε έναν λογικό αριθμό 8 Ιουνίου, το μεσημέρι, 12 η ώρα δηλαδή, θα συζητήσουμε για τις οπολογίες αυτές συμπεριλαμβανομένων και των συμβιβαστικών τροπολογιών που θα συντάξει η εισηγήτρια και θα, διαπραγματευτούν, θα διαπραγματευτεί η εισηγήτρια στις 12 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στις 13 Ιουνίου. Ε, λοιπόν, τελειώσαμε εδώ και θα συζητήσουμε τώρα για, τον, για την εντολή που δίνουμε στον, ε, στην Επιτροπή για, την, για τον Τρίλογο. Εντολή που δίνουμε για τον Τρίλογο για την, με την, ε, και για την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να διευκρινίσω δύο-τρία πράγματα διότι υπάρχουν κάποια προβλήματα νομίζω με αυτό τον κατάλογο ψηφοφοριών. Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Λοιπόν, δεν, για την τροπολογία που, τέσσερα που έχουν υποβάλει οι πράσινοι του κύριου Κάσλερ. Δεν βλέπω εγώ τη χρησιμότητα. Και επειδή δεν θέλω να είμαι και ιδιαίτερα δυσάρεστη, ε, και μου ζητήσανε να γίνει και μια δυνατότητα να υποβάλουν προφορική τροπολογία. Τους δίνω, θα τους δώσω το λόγο ε, να μου πούνε αυτή η προσθήκη, το such as και τα λοιπά, πώς ε, διευκρινίζει περαιτέρω την τροπολογία του κύρου Κάστλερ. Θα ήθελαν, θα ήθελαν οι πράσινοι να το διευκρινίσουν. Yeah. Sorry, they, um, you know, our view was that this we we've shifted Αλλάξαμε λίγο το κόμμα εκεί και το βάλαμε το σατσάς και τα λοιπά, γιατί θεωρούμε ότι με τα παραδείγματα που περιγράφουμε εδώ δεν είναι ότι θέλουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να συμπληρωθούν στην αστυνομική γραμμή, στην αστυνομική, στην αστυνομική γραμμή αυτή, αλλά απλώς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων που να προβλέπεται για, τον, ε, για τη γραμμή αυτού του προπολογισμού. Επομένως, το, στον κατάλογο των, των ψηφοφοριών η τροπολογία δεν αφορά το EG, αλλά ε, αφορά όλο αυτόν τον, κατάλογο των δραστηριοτήτων που περιγράφονται, που ξεκινάνε με το such Η, η τροπολογία, η τωρινή προπολογία αναφέρει παραδείγματα κάποιων δημοσιονομικών γραμμάτων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η τροπολογία μας αυτό το οποίο θέλει είναι να αναφέρει ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας κάποιες ε, δημοσιονομικές γραμμές. Αν θέλετε να ε, αλλάξουμε την σειρά, την επαναδιατυπώσουμε την, την ε, παράγραφο. Αλλά το σάτσα άσα πρέπει να παραμείνει όμως, λέει η κυρία Περές. Ναι, κρατήστε το, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει η κυρία Περές, η... αλλάζει η σειρά της παραγράφου, της πρότασης, αλλά τι θα γίνει με αυτό το IG και το such as, θα τα αφήσουμε, χρειάζονται, δεν χρειάζονται. Κοιτάξτε, εάν τυχόν είναι να δημιουργήσουμε τέτοια, τέτοιο χάος, ας μην το έχουμε, ας μην την κάνουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Καλώς, λέει η κυρία Μπερές, ευχαριστώ για την σύνεση και τη σοφία σας. Ε, παραμένει το κείμενο τροπολογία ως έχει. Τώρα, γκουε, τροπολογία 9, αποσύρθηκε διότι όπως συμφωνήσαμε και χτες, ε, την έχουμε με το στην προφορική τροπολογία, ε, στην τροπολογία 21. Δεν ξέρω τι έγινε. Όπως επίσης ε, σας είχαμε ζητήσει την άποψή σας για την τροπολογία 13. Σας είχαμε ρωτήσει την αποσύρετε ή όχι. Euh, Καλημέρα. Τι διατηρείτε. Πολύ ωραία, εντάξει. Ο Σόρι. Όρη. για το 17 υπάρχει ένα πρόβλημα, όντω στην πρότασή μα. Ε, Είναι προφορική η τροπολογία. Εμείς μιλάμε για union programs. Για τον όρο μετανάστες, μικρό. Αυτό θέλαμε να διαγράψουμε. Και δεν θέλαμε να έχουμε έναν κατάλογο, όχι όπως σαν τους Ρωμά, αλλά να πούμε και μετανάστες διότι ένας κατάλογος, ο οποίος δεν θα είναι εξαντλητικός, θα ανέφερε κάποια άτομα, άτομα συγγνώμη, και θα προκαλούσαμε συζητήσεις, ε, αέναες συζητήσεις, εξού και πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητάμε για ευάλωτες ομάδες. Σας κατάλαβα καλά κύριε Ωρέ, Θέλετε καταρχάς να ψηφίσουμε σε ένα πρώτο μέρος το Stress That the Union Programs Must τα προγράμματα της Ένωσης οφείλουν να προσανατολίζονται σε ευάλωτες ομάδες και όλα τα υπόλοιπα να, να είναι σε, μια δεύτερη ομάδα, σε ένα δεύτερο κομμάτι που θα ψηφιστεί ξεχωριστά. Δηλαδή να μιλήσουμε για μετανάστες όπως η Ρωμά. Αυτό δεύτερο, να είναι δεύτερο κομμάτι. Όμως δεν έχουμε φτάσει εκεί γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα. Υπάρχει τροπολογία 15. Εδώ για την τροπολογία αυτή υπάρχει και μια προφορική τροπολογία η οποία επιβλήθηκε σήμερα. Και εδώ έχουμε δύο δυσκολίες. Το δε, ποια είναι, ότι αν η 15 κάνει να εκπέσει η, 13, η 16, συγγνώμη, η 16 θα ήθελα να προσθεθεί σαν προσθήκη, να προσθεθεί στην τροπολογία 15. Επομένως, η τροπολογία θα λέει γιατί αλλιώς χάνουμε την έννοια της δημιουργίας των ενδιάμεσων περιοχών που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Λοιπόν, η 15 θα λέει τα εξής. Θεωρεί ότι η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ενδιάμεσων περιοχών μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Συνεχής θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αίτημα για αύξηση και μετά διατηρείται το κείμενο ως έχει. Λοιπόν, για αυτή την προφορική τροπολογία σας είχα πει χτες ότι θα γίνει μια ε, διαβούλευση με την εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μας είπε η κυρία Μωρέο ότι δεν ε, συμφωνεί με αυτή την τροπολογία διότι θέλει να αυξηθούν οι πόροι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είχαμε περάσει από το διπλασιασμό σε αύξηση και οφείλω να ε, ομολογήσω ότι ε, με εντυπωσιάζει κάπως, με εκπλήσει η στάση της συζητητριάς μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι αν δούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα από τα καλύτερα ταμεία, χρησιμοποιείται, οι πόροι του χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και όπως είχαμε πει και με τον Επίτροπο, θέλουμε ε, να αυξηθούν τα κονδύλια, να αυξηθούν οι πόροι που ε, αφιερώνονται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε και εμεί σαν Επιτροπή. Επομένως, μέσα στα πλαίσια ε, του, της εντολής που δίνουμε για τον τριμερή διάλογο, θεωρώ ότι είναι παράλογο να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε, ευθύ εξ αρχή οποιαδήποτε ιδέα για ε, διπλασιασμό των πόρων και να μιλάμε μόνο για αύξηση. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι ε, με ενδιαφέρουν ε, πάρα πολύ όλα τα κοινωνικά προγράμματα, όλη η κοινωνική πολιτική που θα βοηθήσει στην ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε όμως, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ε, με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητάμε τα αδύνατα. Και δεν μπορούμε να ζητάμε τον διπλασιασμό Μα δεν μιλάμε για... Να τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν μπορούμε να ζητάμε τον διπλασιασμό των, της ε, πρικοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ε, διότι ούτως ή άλλως με την ε, πρόφαση ότι στα ευρωπαϊκά ταμεία δεν ε, έχουμε διαθέσιμους πόρους ούτως ή άλλως. Ο προπολογισμό δεν μπορεί να διπλασιάσει την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχουμε ένα ποσοστό χρησιμοποίησης αν θέλετε, των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που ανέρχεται στο 82% του, του, ποσού, του συνολικού ποσού που προβλέπεται με μεγάλες ανισότητες. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό τι σημαίνει να ζητάμε και μέτρα ε, μέτρησης του, των συνεπειών, του αντικτύπου και να μην προσανατολισόμαστε σε ενδιάμεσα επίπεδα και να μην ε, είναι προς όφελος των μισθωτών των ιδίων. Επομένως, εάν μια πρώτη απέτηση είναι να αποφελούνται οι μισθωτοί και δεύτερον να ε, μην ε, χρησιμεύει για τους ενδιάμεσους, ήδη θα έχουμε μια αύξηση των πόρων του, των διαθέσιμων πόρων. Δεύτερον, δεν είπα ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι πόροι του κοινωνικού ταμείου, απλώς πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Ευρώπης, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι μπορεί να γίνει και να ξέρουμε τι είναι ανέφικτο. Δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ε, υλοποιηθούν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση θα ήθελα λέει ο κύριος Σέρκας, γιατί η κυρία Μωρέ μιλάει για διπλασιασμό του Ταμείου. Ε, θα κατανοούσα ε, κάτι τέτοιο ως δικαιολογία ε, αν πρόκειται για διπλασιασμό, αλλά η τροπολογία που έχω εγώ δεν μιλάει για διπλασιασμό, μιλάει για αύξηση. Θα ε, με διέφερε ε, να μάθω τι λέει η κυρία Μόρα, γιατί δεν πρόκειται για διαπλασιασμό. Έχει εξαφανιστεί αυτό. Γίνεται πλώς λόγος για αύξηση των πόρων, χωρίς ποσοτικοποίηση. Alors, nous allons euh, passer au vote. Pardon, Madame Morin. Η κυρία για τα, αυτό που λέει ο Αλεχάνδρος Σέρκας. Είναι θέμα στρατηγικής. Αυτό που δεν θέλω εγώ είναι αυξάνοντας την πρικοδότηση του ε- Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να συμπεριληφθεί εκεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Ήταν λάθος αυτή η συγχώνευση. Ε, σε αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας διότι συχνά ακούω να γίνεται λόγος γι' αυτό. Και κανείς από εμά, καμία πολιτική ομάδα δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ξέρω, Αλεχάνδρο, ότι και εσένα σε ενδιαφέρει πολύ, όσο και μένα να γίνεται αυτή η διάκριση και έχουμε και άλλους συναδέλφους που θα το φροντίσουν να υπενθυμίσω στην κυρία Μωρά ότι υπάρχει μία τροπολογία που διευκρινίζει ακριβώς αυτό το σημείο και θα το ψηφίσουμε ούτως ή άλλως. Επομένως, το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να υπάρχει, ε, δεν, να γίνει συγχώνευση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με το Ταμείο Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ΕΛΚ θα πρέπει να πει ότι δεν θέλει αύξηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κύριο Έγγελ. Μία διευκρίνηση κι εγώ. Έχω την ε, αίσθηση ότι σήμερα το απόγευμα η, η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για να συντάξει ομοδότηση του Κοινοβουλίου για τις μεσονομικές προοπτικές θα ψηφίσει να παραμείνει ε, το, Ευρω... το Ταμείο για την Προσαρμογή για την Παγκοσμιοποίηση ως έχει. Επομένως, η ανησυχία σας ε, δεν νομίζω ότι δικαιολογείται μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών όπως είναι τώρα. Επομένως, κανείς δεν επιθυμεί, ή τέλος πάντων μπορεί να το επιθυμούν κάποιοι, αλλά δεν θα είναι η άποψη του Κοινοβουλίου, ε, να μην αυξηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Νομίζω ότι μια τέτοια διατύπωση είναι απόλυτη εφικτή. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Καθυστερήσαμε λίγο. Ε, αλλά, ε, λοιπόν, ε, τροπολογία 1, κυρία Κατά, ε, ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Φιγκερέντο, Λογιαρίκ. Υπέρ κατά, αποχέ, νομίζω εγκρίθηκε, αλλά μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Τέλο πάντων, οι διευκρινήσει που έγιναν προηγουμένω νομίζω ότι ήταν ε, χρήσιμε. Όλοι έχετε τι κάρτε σα, Λοιπόν, όλοι είσαστε οπλισμένοι για να ασκήσετε το δημοκρατικό σα δικαίωμα. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρασε ψηφοφορία. 23 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, συμβαστική πρόταση α, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 4. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 5, προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 6. Παράγραφος 4, συγγνώμη, τροπολογία 6, Φιγκερέιντο Λεγιαρίκα. Με το προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της κυρίας Τούρινεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέχεστε επομένως να ψηφίσουμε την αρχική παράγραφο 4. Κατά τις συνθήκες. Πολύ ωραία. Ψηφίσουμε την παράγραφο 4 στην αρχική της μορφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 8 του κυρίου Ρή. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ίδια διαδικασία, επομένως, πρέπει, μπορούμε να ψηφίσουμε την αρχική παράγραφο 5. Ψηφίζουμε, αρχική παράγραφος 5, υπέρ. Α, δεν χρειάζεται. Υιοθετείτε αυτόματα. Πολύ ωραία. Α, αυτόματα εγκρίνεται, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Θα, θα κρίνεται αργότερα το τρόπο προεδρίας μου. Λοιπόν, θα με βαθμολογήσετε μετά. Ε, Λεγιαρίκα Φιγκερέιντο, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 11, κυρίες Τουρίνεν και κυρίες Κορνίλισεν, υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε ηλεκτρικά. Τροπολογία 11, ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Ψηφίσατε? Πέρας ψηφοφορίες. 24 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται, υιοθετείται. Επομένως, καταπίπτει η τροπολογία 10. Παράγραφο 7. Τροπολογία 12 της κυρίας του Ρίνεν και Σρέτερ των κυρίων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Φιγκερέιντο Λογιαρίκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 7. Τροπολογία 14 των ιδίων υπέρ κατά αποχές θα το εξακριβώσουμε επαλήθευσης, ηλεκτρονική επαλήθευσης. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη 19 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία... Τροπολογία 8 λέει η, η, κυρία Περέσα. Ε, είναι παράγραφος 8, τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Παράγραφος 9, τροπολογία 17 κυρίου Ορή σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ψηφίζουμε χωρίς ε, το Migrants και Ρώμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της προσθήκης των λέξεων μετανάστες και Ρωμά. Υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά καλό να το επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη 18 υπέρ, 24 κατά. Οι προσθήκες αυτές απορρίφθηκαν. Τροπολογία 18 του κύριου Γιωβίνα, που είναι συμβατή υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίσουμε μετά την παράγραφο 9, την τροπολογία 19, Φιγκερέιντο και Γιαρίκ, ε, Γιαρίκ υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 της κυρίας Αρκή είναι υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται, ε, ε υιοθετείται. Ε, τροπολογία 21 με την προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 της κυρίας Τούρινεν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 23 αποσύρθηκε, επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 24 της Ήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25, Γεωβίν και Χαρκίν είναι συμβατή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και μετά την παράγραφο 10 έχουμε την τροπολογία 27 του κυρίου Μπουλόν με μια προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 4 κατά και 0 αποχές. Επομένως, η εντολή μας ε, για τον τρίλογο έχει υιοθετηθεί για τον τριμερή διάλογο. Τώρα, θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση της κυρίας Γκίρλιν για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας στα πλαίσια της νομοθεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις. Παράγραφος ένα... Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 2. Συμβαστική πρόταση α. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 3. Τροπολογία διαγραφή για τη διαγραφή ενό κειμένου. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική πρόταση F. Υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Στην παράγραφο 7 όχι, παράγραφος 4, τροπολογία 7 αποσύρθηκε, επομένως ε, ψηφίζουμε τη συμβασική τροπολογία Β, ε, υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4 έχουμε τροπολογία 12 του Κοφεράτη, με ζητάει ξεχωριστή ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι τώρα, το πρώτο κομμάτι. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου κομματιού που δεν έχει το calls accordingly for them to be increased. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι Κόλς, ακρόλυτη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην παράγραφο 5, τροπολογία 13, απορρίφθηκε, ε, συγγνώμη, αποσύρθηκε. Άρα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία σε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μετά την συμβαστική αυτή ε, πρόταση έχουμε την τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 9, Μετά την παράγραφο 5 έχουμε τη συμβαστική πρόταση ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Κυρία Ρέγνερ. Εξ Ξενόματος των συντακτών της τροπολογίας 8 θα ήθελα να την αποσύρουμε. Λοιπόν, συμβιβαστική πρόταση D. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίδεται. Τροπολογία 24. Όχι, 21 καταπίπτει και η τροπολογία 24 οι τροπολογίες 22-23 Α, ζητώ συγγνώμη. Την 24 πρέπει να την αποσύρουμε. Διότι... Α, όχι. Πρέπει την 24 πρέπει να την ψηφίσουμε. Διότι το δεύτερο κομμάτι της 12 δεν ψηφίστηκε, ενώ η 18 αποσύρθηκε. Επομένως ε, ψηφίζουμε, την τροπολογία 24. Υπέρ. Τη κυρία Φιγκερέιντο. Θέλετε να σας διαβάσω την τροπολογία 24. Επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει ένα γενικό κατόφλι για την ε, πληρωμή των, ε, από, καταβολής, για την καταβολή αποζημιώσεων στους μισθωτούς ε, που θα πρέπει Κατά τι διαδικασίε ελευθερικότητα, αντίστοιχα τουλάχιστον με ένα μήνα μισθού για κάθε έτο εργασία, η καταβολή αυτή πρέπει να διασφαλίζεται άμεσα από το οικείο κράτο μέλο, το οποίο στη συνέχεια θα ζητεί το αντίτιμο κτλ. κτλ. Υπέρ. Για την τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20, ή μάλλον οι τροπολογίες 22, 23, 25 και 26 αποσύρθηκαν. Επομένως, έχουμε την τροπολογία 27 που είναι για να διαγραφεί το κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 7... Ψηφίζουμε την τροπολογία 28 του κυρίου Μπουλό με μία προφορική τροπολογία. Ή έχει κανείς αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Ναι. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 28 όπως ήταν αρχικά. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 28 χωρίς την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 καταπίπτει. Επομένως, στην παράγραφο 8 ψηφίζουμε την τροπολογία 30 της κυρίας Ρέγνερ και άλλων. Ε, ζητάνε να διαγραφεί το κείμενο υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Je peux pas changer mon vote. Ah, si. Ε, tout le monde a pu voter Le vote est clos. 21 υπέρ, 21 κατά και 2 αποχές. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 20, 31 του κ. Μπουλόν. Υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά καλό θα είναι να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 31. Tout le monde a pu Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 14 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Επομένως οι τροπολογίες 32-33 καταπίπτουν. Μετά έχουμε την τροπολογία 34 του κυρίου Κοφεράτη σε δύο κομμάτια. Ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι χωρίς το and considered μέχρι το non-standard contracts. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ποιος ε, είναι υπέρ της προστίκης ε, του δεύτερου κομματιού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 9, τροπολογία 35 του κυρίου Μπουλό, σε δύο κομμάτια, σε δύο τμήματα. Ε, με μια γλωσσική παρατήρηση για το αγγλικό, την αγγλική εκδοχή. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, χωρίς δηλαδή end with threshold levels κτλ. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο κομμάτι τώρα, την προσθήκη των λέξεων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9 έχουμε τροπολογία 36 της κυρίας Γκίρλινγκ με μία προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 της κυρίας Ρέγνερ με μία προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, υιοθετείται. Μετά την παραγράφο 9 έχουμε τροπολογία 38 της κυρίας Ρέγνερ υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 39 του κυρίου Μπουλόν υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 30 Ρέγνερ υπέρ κατά. Ε, συγγνώμη 40 υπέρ κατά αποχέ. Μετά τροπολογία του κύριου Κοφεράτη 41 υπέρ κατά ε, υιοθετείται. Ε, τροπολογία 42 Ρέγνερ με μια προφορική τροπολογία και ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία. Αν όχι, ψηφίζουμε το, κομμά... το κείμενο σε δύο τμήματα. Το πρώτο κομμάτι χωρί το the additional μέχρι το proceedings. Υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται για την προσθήκη τώρα των λέξεων δεύτερο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές θα το επαληθεύσουμε. Le vote est ouvert. ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι υπέρ. 23 ψήφοι υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Η 43-44 αποσύρθηκε. Μετά την παράγραφο 9 ψηφίζουμε την τροπολογία 45 του κυρίου Μπουλό με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 μπουλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 αποσύρθηκε. Ψηφίσουμε την τροπολογία 48 του κ. μπουλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 49 της εισηγήτριας με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνθηκε. Άρα ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ε, ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 33 ε, υπέρ, 3 κατά, 8 αποχές. Συγχαίρουμε την εισηγήτριά μας. Nous en avons terminé avec notre Πάνε ψηφοφορίες. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αντάμ Κάσα, ε, εισηγητή για το σημείο 19, για να εξτάσουμε τις τροπολογίες στην έκθεσή του με θέμα κινητικότητα και ένταξη ατόμων με αναπηρίες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Να περιμένουμε δύο λεπτά να καταλαγιάσουν τα πνεύματα λίγο. Ε, λοιπόν, παρακαλώ να διακόψετε τις ιδιωτικές συζητήσεις και τα υπόλοιπα πηγαδάκια για να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε. 298 τροπολογίες έχουμε συνολικά κάνει και εγώ πολλές για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη δομή και τη διάρθρωση της έκθεσής μας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Νομίζω συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Χαίρομαι για τις περισσότερες από αυτές. Προσθέτουν πραγματικά και βελτιώνουν το κείμενο. Το είπα και στην πρώτη συζήτηση και θα ήθελα να το επαναλάβω και σήμερα. Μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη συνένεση στις πολιτικές ομάδες ε, υπέρ των ατόμων με αναπηρία. Φαίνεται και από τις τροπολογίες 298 σας είπα κατατέθηκαν. Δεν είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω όλους σας ε, και για τις 298. Ε, Καταλήξαμε όμως σε 21 συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν το 1 τρίτο των κατατεθήσεων. Ε, μεσολάβησε και η γαλάζια εβδομάδα, η ε, τυρκουάζ, και αυτό δεν μπόρεσα να δω όλους τους συντάκτες. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να το κάνω. Έχουμε και άλλες ε, γνωμοδοτούσεις επιτροπές, δύο. Σήμερα θα ψηφίσει η τρίτη και είμαι πεπισμένος ότι και οι γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών θα ενταχθούν στην έκθεση. Με χαρά θα το προτείνω κι εγώ. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω μερικά ζητήματα ε, για να ακούσω και την ε, άποψή σας. Δεν θέλω να γίνει συζήτηση για την παράθεση, αλλά από κοινού να σκεφτούμε πώς θέλουμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Το ίδιο ισχύει και με τη συνέχεια που δίνεται ε, και παρακολούθηση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν γίνει και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόμα δεν έχουμε αποκρισταλωμένη άποψη, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έχει κάνει προτάσεις και το φόρουμ των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να υπάρξει λοιπόν μια επιτροπή που να εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις. Ε, Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφες οι στατηγικές ε, με τις ίδιες έννοιες, να μετρούν τα ίδια στοιχεία δηλαδή. Όπως και στην προηγούμενη συζήτηση, σε αυτό το κείμενο ε, μας απασχολεί το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Έχουν γίνει πολλές τροπολογίες και προς τα δω. Νομίζω επιβαρύνουν κάπως και περιπλέκουν το κείμενο οι τροπολογίες αυτές. Χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση, επαναλαμβάνω. Ε, για κάποιες ειδικέ κάρτες ή διαβατήρια, μια κάρτα κινητικότητας ατόμων με αναπηρία, ένα πάσο, δεν ξέρω κάτι, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις τους τα άτομα με αναπηρία. Μια ταυτότητα ε, θα το συστήσω με του πιο δεν χρειάζονται υπερβολές εδώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ε, σε όλα τα κρατη και αυτού του είδους οι κάρτες, οι ταυτότητες ε, ατόμων με αναπηρία βοηθούν. Επίσης, ε, έγιναν πολλές τροπολογίες για αγαθά και υπηρεσίες. Πώς θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση δηλαδή τα άτομα με αναπηρία σε αυτά στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Δύο είναι οι τροπολογίες που ασχολούνται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείε εκείνες που προσλαμβάνουν περισσότερο άτομα με αναπηρία από όλες τις επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο και καλά κάνουν και το λέμε και στις τροπολογίες για τη στρατηγική του 2020 επίσης χαιρόμαστε. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης. Άλλο θέμα που αναφέρουν οι τροπολογίες και χρειάζεται η συμβιβαστική πρόταση είναι το εξής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τις διοικήσεις, ε, τις δημόσιες διοικήσεις δηλαδή, τον κρατικό μηχανισμό για να ε, διαχειρίζεται τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Τα έγγραφα, πόσα είναι πιο προσβάσιμα, η ενημέρωση, η πληροφόρηση, γενικότερα. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των παιδιών με αναπηρία. Πώς θα γίνεται η συνεργασία με τους γονείς τους. Όλες οι τροπολογίες ασχολούνται με το θέμα αυτό από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία προσέγγιση προς την κατεύθυνση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Στα κράτη-μέλη φαίνεται δεν το έχουν καταλάβει ακόμα αυτό και εμείς αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η κύρωση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάποιου παραρτήματος που έχει εθελοντική ισχύ και όχι δεσμευτική ε, πρέπει να μας απασχολήσει και να παρακολουθούμε την εφαρμογή για την επόμενη δεκαετία. Έρχομαι τώρα στα δημόσια έργα και τις κρατικές ε, προμήθειες έχει γίνει πρόταση να ε, διευκολυνθεί η πρόσβασή τους. Να υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία και γενικότερα συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Είναι μεγάλη η λίστα, μακρύς ο κατάλογος. Ε, έρχομαι τώρα στα συγκεκριμένα μέτρα. Όλα αυτά που προτείνουν οι συνάδελφοι δεν μπορώ παρά να τα υποστηρίξω διότι έχω την εντύπωση ότι αυτή η έκθεση μπορεί να είναι έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά για να πετύχει υπάρχει μια προϋπόθεση. Να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάτι που ακούστηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια ρεαλιστική έκθεση, όχι ένα ευχολόγιο, ε, μια αναλυτική απαρίθμηση καλών προθέσεων. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα που να εφαρμόζονται. Ε, να είμαστε δηλαδή στην πραγματικότητα, στα απτά, στα χειροπιαστά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν έχουν χώρο εδώ στις ε, τροπολογίες και δεν θα τις υποστηρίξω. Ας πούμε, ε, κατώτατος μισθός. Αυτό τι σχέση έχει με τα άτομα με αναπηρία. Δεν ε, εμπίπτει στο πεδίο αυτή της έκθεση να ασχολούμαστε με θέματα κατώτατου του μισθού. Άλλο θέμα. Να γίνει, λέει, ταξινόμηση, ιεράρχηση των ε, υπηρεσιών. Και πάλι δεν έχει θέση ε, αυτή η πρόταση στην έκθεση Πώς, γιατί να τις ιεραρχήσουμε, να τις ταξινομήσουμε. Όλα τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι, οι πάντες θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, χωρίς καμία ε, ταξινόμηση αυτών, ούτε η ιεράρχηση τους. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζονται και οι δραστηριότητες των ατόμων με αναπηρία. Ε, είναι μια επένδυση σε αυτούς για να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, να είναι ισότιμοι πολίτες και φορολογούμενοι που θα συνεισφέρουν στο γενικότερο καλό. Ευχαριστώ για τις 298 τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε. Αυτό δείχνει τι σημασία δίνουν οι συνάδελφοι στην έκθεσή σας. Κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Δεν τα κατάφερα να υποβάλω τι απολογίε που ήθελα, γιατί απουσίαζα λόγω τη προθεσμία, ε, κατά την λήξη τη προθεσμία. Πάντω είμαι και για την εθνική task force που αναφέρατε. Τι εννοείται ανεξάρτητους φορείς ε, πολιτικής που ήδη έχουν ε, δημιουργηθεί υπάρχει η Επιτροπή Ισότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Quality Commission. Ε, εννοείται κάτι τέτοιο εθνική task force, ομάδα δράσης ή εννοείται την καλύτερη υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την Επιτροπή Αναπηριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία επί της αρχής, αλλά το θέμα είναι πώς ακριβώς θα λειτουργεί, πώς το βλέπετε στην πράξη να οργανώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια-δυο αιτήσει για τροπολογίε από άλλου συναδέλφου. Την τροπολογία 49 για τα ωφέληματα από τι αναπηρίε. Εδώ, για τα επιδόματα των αναπηριών. Εδώ θέλουμε κάποιε διευκρινήσει. Δεν είμαι βέβαιη ότι καταλαβαίνω ακριβώ το νόημα. Στην 2.39. Ω ελεύθερη Ουδέποτε είμαστε υπέρ τη ε, αντιστάθμισης και τη αποζημίωσης, των ευθύνων αποζημίωσης, ε, τη υποχρεωτική. Θα πρέπει να είναι σε θελούσια βάση αυτά και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εξακολουθήσουμε και στην ψηφοφορία. Για την οδηγία κατά της διακριτική ε, μεταχείρισης και την τροπολογία 278 για το πώ θα πρέπει να ε, προωθήσει το Συμβούλιο τελικά ε, την ε, οδηγία για τις αναπηρίες και την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα εμπορεύματα. Σίγουρα πρέπει να προστατευτούν εδώ δικαιώματα των αναπήρων. Όμως η οδηγία υπάρχει, κάποια κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει μπλόκο για, την, για να περάσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και θα πρέπει να το υπερβούμε το εμπόδιο. Διότι Εάν δεν θέλουμε διακριτική μεταχείριση στην απασχόληση, δεν θέλουμε το ίδιο ούτε στην πρόσβαση στα αγαθά και τι υπηρεσίε. Η οδηγία αυτή νομίζω θα απελευθέρωνε πολλά. Θα μπορούσε να άρει πολλούς από του φραγμούς που προβάλλονται στους ε, αναπήρους. Εδώ, τώρα στις αναφορές μα για του αναπήρους, μπορούμε να είμαστε συνεπεί σε όλη, σε όλη την έκταση της έκθεσης να λέμε άνθρωποι με αναπηρίες ή ανάπηρα άτομα. Να αναφέρεται όρος people, να μην δίνεται έμφαση στην αναπηρία αυτή καθεαυτή. Και στην τροπολογία 20 προκύπτει αυτό το πρόβλημα και αλλού. Ίσως είναι θέμα μετάφρασης, επειδή μεταφράστηκε από άλλη γλώσσα προς τα αγγλικά. Αλλού λέγεται the disabled στα αγγλικά και αλλού λέγεται disabled people. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε συναπεί και στη διερμηνία το ίδιο και στι ερμηνείε μας. Στην 60 τώρα. τίνεται να κάνετε μία διαφοροποίηση μεταξύ του ιππίου και του μετροπαθούς. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε τέτοια διάκριση. Ποιος θα αποφασίσει ποιες είναι οι ελαφριές ή ήπιες μορφές αναπηρίας οι μετριασμένες και για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει αυτό να είναι ένα κριτήριο. Νομίζω ότι πάμε πολύ μακριά προσπαθώντας να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να έχουμε από την αρχή καθορίσει σωστές ε, αρχές ω βάση εργασία για να τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Αλλά αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε πολύ μακριά σε ορισμούς που κανείς δεν θα ξέρει πώ να του υλοποιήσει σε επίπεδο κάτου μέλου, εκεί θα δημιουργηθούν προβλήματα. Όμω, είναι βέβαιο ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά, όπω έχουμε κάνει και στο παρελθόν, για τα δικαιώματα των αναπήρων και τα θέματα του και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα μα ε, επιτρέψει πάλι μια πολύ καλή μορφή συνεργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Α, ας έφυγε ο κύριος ο κύριος Μάν, δεν Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και σένα, Άνταμ. Πάρα πολύ καλή έκθεσή σου, εξαίρετη. Και γι' αυτό και δώσει τροπολογίες. Το ζούμε όλοι. Σε πολλά κράτη-μέλη τα άτομα με αναπηρίες υφίστανται διακρίσεις, δεν λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις ε, προς ε, την κατεύθυνσή τους και πραγματικά η δική σου προσέγγιση είναι αυτό που χρειαζόμαστε η έκθεση αυτή βέβαια είναι μόνο έκθεση πρωτοβουλίας. Αλλά δεν θα πρέπει να καταντήσει όπως πολλές άλλες εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας κάποια στιγμή Δευτέρα βράδυ να ψηφιστεί περίπου εμπιστευτικά στο Στρασβούργο και να μην το πάρει κανείς είδηση. Να είναι σημαντικό το θέμα. Να δοθεί η σου σημασία. Ε, έχεις δίκιο που λες ότι χρειαζόμαστε ενιαίες στατιστικές γνωρίζω ότι πολλές φορές λένε τα κράτη-μέλη «Ε, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε όλα αυτά που κάνουμε. Όχι, να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Ε, διατηρούν την αυτονομία τους τα κράτη-μέλη, αλλά να ε, είναι παρόμοιες οι στρατηγικές για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να έχουμε ένα γνώμονα για την αξιολόγηση. Η 284 δική σου τροπολογία εξαιρετική συνδέεις εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Ακριβώς οι ε, άνθρωποι με αναπηρίες στην Ήπεθρο αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι αλλού. Γι' αυτό χρειάζεται σύνδεση και να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως έχουν στοιχεία να μας βοηθήσουν. Πολύ σημαντικό αυτό που ζητάς. Επιτρέψε μου να αναφερθώ στη δική μου τροπολογία υπαριθμό 48 που δεν το έχουν ζητήσει άλλοι συνάδελφοι είναι οι γυναίκες με αναπηρία που υφίστανται διπλή διάκριση. Έχουμε τώρα και το gender mainstreaming και τη διάσταση του φύλου δηλαδή σε όλες τις πολιτικές και θα πρέπει να το φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής, όχι στο περιθώριο. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί η τροπολογία 48 με αυτή τη διατύπωση. Είπε ότι θέλεις να συζητήσει μαζί μας συμβιβαστικές προτάσεις, πολύ σημαντικό. Και επίσης συμφωνώ με τη Λίζ Λίν για την κοινωνική ευθύνη των εταιριών και ο κύριος Κοφεράτη στη 239 ζήτησε να είναι δεσμευτικό, να είναι υποχρεωτικό. Όχι, εγώ δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί. Να διατηρηθεί η πίεση για την κοινωνική ευθύνη των εταιριών, όχι όμω υποχρεωτικό. Να παραμείνει σε εθελούσια βάση. Ορισμένε επιχειρήσει το πράττουν θαυμάσια, άλλε κρατούν ακόμα αποστάσει. Θα πρέπει να τους πούμε όμως ότι έχουν και εκείνοι κοινωνική ευθύνη. Αλλιώ πώ θα γίνει αποδεκτή αυτή η έννοια τη κοινωνική οικονομία τη αγορά που έχουμε στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με τους ηγητέ και του υπολείπου, νομίζω ε, θα πάνε καλά τα πράγματα όπως μας έχει συνηθίσει πάντα με πνεύμα συνεργασίας και τελικά μια έκθεση που θα είναι μια σημαντική φωνή. Έχει δίκιο η Λίν και για την ορολογία. Είναι άτομα με αναπηρία, δεν είναι ανάπηροι. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να το λέμε. Ε, η κυρία και μετά η κυρία Η συνάδελφος Μπλίνκεβιτσούτε αυτή τη στιγμή ε, είναι στην Επιτροπή Ελευθεριών σε ψηφοφορία. Ε, κολλιέται. Θα συνεχίσω εγώ στα αγγλικά να σας πω αυτά που μου έδωσε να σας διαβάσω. Υποστηρίζω τις τροπολογίες αυτές γιατί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που ε, έχουν ακόμα ε, ε, στην Ευρώπη τα άτομα με αναπηρία είναι μεγάλη ανεργία. Δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να πηγαίνουν σε σχολεία ή σε χώρους κατάρτισης γιατί δεν έχουν ειδικά προγράμματα για αυτούς. Επίση δεν υπάρχουν ε, κατάλληλοι επαγγελματίε και επίση τα σχολεία ε, δεν ε, έχουν τη φυσική πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Στη συνέχεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια ε, της ελεύθερης έκφρασης των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε εκλογές. Μικρό μόνο ποσοστό ατόμων με αναπηρία συμμετέχει σε εκλογές γιατί δεν είναι εύκολη η πρόσβαση ε, στα εκλογικά τμήματα, δεν είναι ε, σύμφωνη με τις ανάγκες τους. Επίσης, ε, πρέπει τα κράτη-μέλη να εθαριθούν, να ορίσουν την αναπηρία και να μην θεωρούν ότι είναι μόνο μία σωματική διαταραχή, αλλά η δυσλειτουργία, αλλά ότι έχει και κοινωνικές προεκτάξεις. Και επίσης η σημαντική τροπολογία αναφέρεται ε, σε, στη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα με πνευματική αναπηρία που ε, είναι πολύ συχνά εκτεθειμένη σε βία και κατάχρηση. Θα πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα δικαιώματά τους, τα ιδρύματα στα οποία είναι έγκλειστοι και θα πρέπει να περάσει η περίθαλψη ε, και στην ψυχική ιδεία από την ιδρυματοποίηση στην κοινωνικοποίηση. Αυτά. Και θα είναι σε επαφή με τον εισηγητή για να συνεργαστούν στο τέλος. Ευχαριστώ. Η κυρία Μωρά και μετά η κυρία Φιγκρέιβο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κώσα για το έργο του. Εγώ η ίδια είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Γυναικών και εργαστήκαμε έτσι ώστε η έκθεση η δική μας να συντονιστεί με αυτήν. Το πρώτο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ είναι ότι Πρέπει πράγματι να αγωνιστούμε για να εξαλείψουμε κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης παρά τις ε, εθνικές πολιτικές που επαγγέλλονται την ε, ένταξη των ε, αναπήρων, των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό το επαγγέλλονται μένα, αλλά δεν το πράττουν. Έτσι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή όλων στην υλοποίηση, την πρακτική εφαρμογή. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ευνοήσουμε την υλοποίηση των πολιτικών με τα νομοθετικά μέτρα που προβλέπονται για τα άτομα που υποφέρουν από κάποια αναπηρία. Εδώ θα συμφωνήσω επίσης σε δεύτερη φάση με τον συνάδελφο Τόμας Μαν, ε, που λέει πρέπει να ρηγονωθεί μια ουσιαστική συζήτηση στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια μια από τις συνόδους. Διότι αν κοιτάξουμε πόσε είναι τροπολογίες και πώς το θέμα αυτό μας κινητοποίησε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Γυναικών. Έχουμε σχεδόν 350 τροπολογίες συνολικά. Άρα μεγάλη, ευρύτατη συμμετοχή και διάθεση και των μεν και των δε να επενδύσουν ε, πολλά στην πολιτική αυτή για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Θα πρέπει λοιπόν να φοβιερώσουμε μια συζήτηση στο σημαντικότατο αυτό θέμα. Τρίτη παρατήρηση, ειδικότερα για τις γυναίκες. Άκουσα τον Τόμας Μαν και διάβασα την τροπολογία 48 που υπέβαλε ο Τόμας. Θα πρέπει να πω ότι αυτός ο άξονας ε, πραγματικά μας ε, οδήγησε και στην Επιτροπή Γυναικών σε μια συγκεκριμένη πορεία. Μιλάμε για διπλή αναπηρία σε κάποιες περιπτώσεις των γυναικών που υποφέρουν από αναπηρία και έτσι επιβαρύνονται με περαιτέρω παράγοντες αποκλεισμού και δυσχεριών στην ε, κοινωνία. Τον ε, καθησυχάζω λοιπόν τον Τόμας Μαν και του λέω ότι ακριβώς το θέμα αυτό το καλύπτουμε πλήρως στην έκθεση της Επιτροπής Γυναικών. Θα ψηφιστεί μάλιστα το απόγευμα. Τέλος, εγώ ίδια πρότεινα τα άτομα που κινητοποιούνται υπέρ της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες να τη χάνουν κάποιες αναγνώρισης σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχει κάποια κύρωση της πείρας τους, των δεξιοτήτων αυτών που ακριβώς θα τον στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. σε πολλές περιπτώσεις, χάρη στην εθελοντική τους εργασία και την προσωπική τους αφοσίωση, καλύπτουν τα όσα δεν πράττει η ίδια η κοινωνία και τα κράτη-μέλη. Άρα δίκαιο το βρίσκω να υπάρχει και κάποια ανταπόδοση, κάποια αναγνώριση της προσπάθειάς τους από την πλευρά των κρατών μελών. Αυτό θα προταθεί και στην ψηφοφορία μας σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Κωσά. Η κυρία Σρέτερ και μετά ο κύριος Γκουτιέρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, σε γενικές γραμμές να θυμίσω μερικά και να συμπληρώσω κάποια άλλα. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Και το θέμα του φίλου μας ενδιαφέρει και μας έχουμε κάνει και σχετική τροπολογία αλλά επειδή είναι τόσο καλή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών, να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες διατυπώσεις και αυτές να υιοθετήσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε η Λίς Λίν για την οδηγία κατά των διακρίσεων. Είναι σημαντικό αυτό το κείμενο ε, για να ε, εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο αυτά τα θέματα. Το ζω καθημερινά ε, πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη απώλεια είναι η μη εφαρμογή τους. Με την οδηγία κατά το διακρίσεων το Κοινοβούλιο τότε είχε ε, παρουσιάσει ένα κείμενο πάρα πολύ ισορροπημένο και πάρα πολύ καλό. Και προέρχομαι από μια χώρα η οποία πρωτοστατεί στην εμπλοκή στο Συμβούλιο, στο συνασπισμό εκεί και μπορώ να διαβεβαίωσω στους αδέλφους από τη Γαλλία και την Αγγλία ότι είναι μόνιμο μέλημά μου σε όλες τις συζητήσεις και στην εκλογική μου περιφέρεια. Προσπαθώ πάντα να οδηγήσω σε απεμπλοκή αυτή την κατάσταση όσο μπορώ. Νομίζω ότι λίγο έχουμε προχωρήσει γιατί πλέον ε, στη Γερμανία επικρατούν άλλες πολιτικές ε, καταστάσεις και συσχετισμοί. Θα ήθελα να έρθω σε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα που είναι η ταυτότητα, και η κάρτα δηλαδή και ο ορισμός. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλουμε όλα στο ίδιο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί συνδέονται συχνά αυτές οι ταυτότητες αναπήρων με ε, τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης και τέτοια και είναι επίμαχο το θέμα. Ε, καλό είναι να έχουν ένα πάσο ας πούμε για τις συγκοινωνίες ε, αυτό εντάξει, αλλά ε, και να λυθεί γρήγορα για να μπορούν να κυκλοφορούν ε, πιο εύκολα και αμοιβαία αναγνώριση, αλλά απόλυτη εναρμόνιση των ταυτοτήτων, των καρτών αναπήρων, δεν νομίζω, γιατί στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικές. Καλύτερα να περάσουμε από την 883 του 2004 για την αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό πρόκειται κυρίως για μη εμφανίσει, μη ορατές αναπηρίες. Και να υπάρχει ένας τρόπος που να ανταποκρίνεται στα ήθη και στις συνήθειες ενός κράτους να τον αγνωρίζουν τα άλλα χωρίς να είναι υποχρεωμένα να το υιοθετούν πάντοτε γιατί υπάρχουν και κοινωνικά επιδόματα στα κράτη-μέλη που συνδέονται με συγκεκριμένες ταυτότητες, με συγκεκριμένες κάρτες και δεν είναι εύκολο να εναρμονιστεί και σε περίπτωση εναρμόνισης γίνεται αυτή προς τα κάτω. Οπότε, δεν θα ζητούσα πολύ μεγάλη ε, ομοιογενοποίηση, είναι αντιπαραγωγική αυτή. Αυτά τα σημαντικότερα, κατά τα άλλα, περιμένουμε χαρά τις συμβαστικές τροπολογίες και διαπραγματεύσεις και θα επιθυμούσα να ενισχυθεί η έκθεση πρωτοβουλίας με τις τροπολογίες, αλλά έχουμε και το θέμα του όγκου ή της έκτασης. Το ξέρει και ο Άνταμ Κώσα ότι υπάρχει ένας περιορισμός χαρακτήρων, όχι λέξεων. Και γι' αυτό ε, συμπληρώνεται από τροπολογίες, τις οποίες έχουμε εκπονήσει Νομίζω η έκθεση θα είναι καλή τελικά και χρήσιμη και σημαντική. Και θα την υποστηρίξουν οι συνάδελφοι και στο μέλλον. Στην Ολομέλεια. Ο κύριος Γκουτιέρης. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση πρώτα απ' όλα. Είναι σημαντική έκθεση αυτή. είναι καινοτόμο αυτό το στοιχείο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συζητήσαμε για τέτοια στρατηγική εγκάρσια και ειδική για τις πολιτικές που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία τα τελευταία χρόνια ε, προχώρησε η ευρωπαϊκή πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μεγαλύτερη φιλοδοξία αν μη τι άλλο ε, στα θέματα των ατόμων με αναπηρίων. Απόδειξη είναι αυτή η πρώτη στρατηγική και η ε, πρόταση που έγινε πριν από λίγους μήνες για να οριστεί ε, η ε, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα που έχει την καλύτερη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ο των τροπολογιών δεν σημαίνει ότι έχει ελλείψεις. Ε, το αντίθετο δείχνει τη φιλοδοξία και το ενδιαφέρον που έχουμε και πώς θέλουμε να βοηθήσουμε να ε, στηθούν αυτές οι πολιτικές με ένα βασικό στόχο και κοινό παρανομαστή που είναι η ισότητα ευκαιριών σε όλες ε, τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρίες και σε σχέση με ε, τους υπολείπους που δεν έχουν καμία αναπηρία. Από την εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, ψυχαγωγία, αθλητισμό, κινητικότητα και τελικά πρόσβαση σε μια ουσιαστική δημοκρατία. Ακούστηκε προηγουμένως και θα ήθελα να το τονίσω κι εγώ το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το πεδίο ε, εκεί για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση. Από κράτος σε κράτος της Ένωσης διαφέρει η κατάσταση και η προσέγγιση για τις πολιτικές αυτές, για την ένταξη την αγορά εργασίας και στις μικρομεσαίες ατόμων με αναπηρίες και θυμίζω ότι πάνω από 80% της απασχόλησης που δημιουργείται στην Ένωση είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Για ε, ενεργές πολιτικές απασχόλησης, για ένταξη στον εργασιακό βίο ατόμων με αναπηρία, γιατί αυτό είναι το πρώτο αίτημά τους όταν μιλάμε με άτομα με αναπηρίες, είναι τι μπορούν να κάνουν, τους ρωτάμε τι μπορεί να κάνει το κράτος για σας, το πρώτο που μας ζητάνε είναι ένταξη στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη φιλοδοξία στις πολιτικές αυτές, ε, αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να έχουν και επιτυχία. Και να μην έχουμε και διπλές διακρίσεις. Έγινε λόγος για τις γυναίκες προηγουμένως που υφίστανται διπλή διάκριση οι γυναίκες με αναπηρία. Επίσης εγώ ανησυχώ όχι μόνο για το θέμα του φύλου, αλλά και η διάκριση των ατόμων με αναπηρία στην Ήπεθρο. Γιατί και εκεί υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που ζουν στην πόλη και σε εκείνους που ζουν στην Ήπεθρο. Γιατί δεν έχουν προφανώς τις ίδιες ευκαιρίες. Επιπλέον πρόβλημα λοιπόν και αδυναμία. Υπάρχουν προβλήματα εκεί, γνωρίζετε, δημοσίων υπηρεσιών, πρόσβασης υποδομών και εξού και η διπλή διάκριση. Άλλες ευκαιρίες έχουν τα άτομα με αναπηρία που ζουν στην πόλη και άλλες εκείνα που ζουν στην Ήπεθρο. Αναγνώριση λοιπόν των συστημάτων, ομιγενοποίηση αν θέλετε των κοινωνικών συστημάτων και ε, να ε, ε, χτιστεί αυτός ο τέταρτος πυλώνας του κράτους πρόνοιας που είναι η ε, φροντίδα εξαρτημένων ατόμων. Υπάρχουν άτομα με διάφορες αναπηρίες και η βοήθεια που χρειάζονται δεν είναι πάντα ίδια. Ε, ούτε η φροντίδα, ούτε η παροχή ε, προστασίας. Πέρα λοιπόν από την παιδεία, την υγεία και το κράτος πρόνοιας υπάρχει αυτός ο τέταρτος πυλώνας που είναι η ε, παροχή φροντίδας στα άτομα με αναπηρία. Κάποιος με ρώτησε τι σημαίνει αυτή η τροπολογία 49 η δική μου αυτό που σας λέω. Υπάρχει τροπολογία 19. Συγγνώμη, 49. Ε, στην αιτιολογική σκέψη ή τα α νέα, μας είπαν τα άτομα με αναπηρίες ότι υπάρχει εξής φόβος. Σε πολλά κρατημέλη υπάρχει μια βαθιά ε, ε, διάσταση ανάμεσα στα αναπηρικά επιδόματα και στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, όταν βρίσκουν δουλειά, τους κόβουν το αναπηρικό επίδομα, που όμως πολλές φορές τους χρειάζεται για να επιβιώσουν, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, γιατί δεν τους φτάνει το εισόδημα ε, που παίρνουν από την εργασία τους. Και πολλές φορές ε, βρίσκονται μπροστά σε ένα εκβιαστικό δίλημα. Ή θα διατηρήσουν το επίδομα ή θα δεχτούν τη θέση εργασία. Ε, κάπως πρέπει να είναι συμπληρωματικές αυτές οι πολιτικές και όχι αντίπαλες μεταξύ τους. Θα πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση και καμιά φορά αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας προκειμένου να μην χάσουν το επίδομά τους. Και πολλές φορές οι πολιτικοί είναι και θέμα κινήσεων, χειρονομιών, ε, συμβόλων. Υπάρχει και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να το πράξουν, γιατί ε, στην πολιτική η χρόνη είναι πιο σημαντική από ό,τι στη γραμματική και η δράση ε, θα πρέπει ε, να είναι κοινή με κοινούς ε, νόμους, αμοιβαία αναγνώριση και εγγύηση, αν μη τι άλλο, σε όλα τα κρατημέλη στη δημόσια διοίκηση να αναγνωρίζεται και όποιος χρειάζεται, ας πούμε, τη νοηματική γλώσσα να έχει πρόσβαση σε αυτή κτλ. Ευχαριστώ πολύ για τελείωσα. Ωραία. Ολοκληρώσαμε ε, με όλους τους ομιλητές και ξαναδίνω τον λόγο στον ε, εισηγητή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ για τους συναδέλφους, για τις παρεμβάσεις τους. Τις άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη μου όλα όσα ακούστηκαν. Ούτως ή άλλως θα υπάρξουν συμβαστικές προτάσεις. Θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε με όλες ε, τις πολιτικές ομάδες να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες να ικανοποιούν όλους. Καταρχάς, να απαντήσω σε αυτά που είπε η κυρία Λίν Αναφερθήκατε σε, σε ένα παράδειγμα στα αγγλικά ε, για τους, σε σχέση με τους ανάπηρους και, τις, και τα άτομα με αναπηρίες, ότι θα έπρεπε να ε, τονίσουμε ότι πρόκειται για άτομα, κυρίως για άτομα, τα οποία έχουν και αναπηρίες. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο προτείνατε είναι ένα καλό μοντέλο, το οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε, διότι ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο Υπάρχουν ε, πολλές ε, οδηγίες οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω ενός και μόνο νόμου. Και αυτή είναι πολύ καλή πρόταση, πιστεύω, η συμβαστική σας πρόταση. Επίσης, υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα πρόταση για την για, τα λιγότερο, για τις λιγότερο ή ε, περισσότερο σημαντικές αναπηρίες. Η περισσοτερο σημαντικες τονίζει ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι λειτουργικές. Και στην αγορά εργασίας και η δική μου εμπειρία δείχνει ότι τα πράγματα ε, δεν είναι και τόσο καλά. Δηλαδή οι εργοδότες ε, βρίσκουν διάφορα παραθυράκια και προσπαθούν να ε, ξεφύγουν. Γι' αυτό οι δύο αυτές κατηγορίες, Mind and Multiple, ήταν πολύ χρήσιμες για, τους, για, τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Και Προφανώς υπάρχουν πάρα πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν ε, ιδιαίτερα σοβαρά, ε, σοβαρές αναπηρίες. Και εδώ δεν μιλάμε να... Δεν, δεν, δεν μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, αλλά μιλάμε για υπηρεσίες που, που παρέχονται σε όλους. Προσπάθησα και εγώ ε, στα αγγλικά να συζητήσω λίγο τα θέματα με τον σκιώδη εισηγητή και διατυπώναμε ούτως ή άλλως τις τροπολογίες και στα αγγλικά. Ε, και ο τίτλος ε, είναι λάθος, διότι δεν μιλάμε για ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Μιλάμε, ενώ τα αγγλικά μιλάει για ένταξη, το inclusion και όχι integration είναι, έχουν διαφορετικές ε, έννοιες ε, ε, οι δύο αυτές λέξεις. Ο κύριος Μαν αναφέρθηκε στις γυναίκες. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με τα θέματα αυτά. Εγώ θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις τους γιατί είναι πάρα πολύ καλές, θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη μου κατά 100%. Μιλάμε για γυναίκες που έχουν αναπηρίες και για γυναίκες που είναι μητέρες παιδιών με αναπηρίες και για τις δύο κατηγορίες θα ε, κάνουμε, θα ε, προσπαθήσουμε να εντάξουμε και τις δύο κατηγορίες. και μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. 80-90 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τις κάρτες, συμφωνώ με τους ομιλητές, τους συναδέλφους. Στην εισαγωγή μου είχα πει ότι θα ήθελα να υπάρξει μια ισορροπία στα θέματα των καρτών για να μην υπάρχουν υπερβολές και αντιρρήσεις. Και νομίζω ότι η συμβαστική μου πρόταση θα απαντήσει και θα καθυσυχάσει τις ανησυχίες. Ο κύριος Πριέτο επίσης εξέφρασε κάποιες ε, ανησυχίες του. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας, θα πρέπει να τα δούμε και κάπως ευρύτερα. Επίσης, σας είπα ότι θα υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες, τις οποίες δεν θα υποστηρίξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι κρίνω οι τροπολογίες αυτές δεν είναι καλές, αλλά απλώς θα ήθελα να αποφύγω να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να, να εκφράσουμε ένα μεγάλο κατάλογο ευχών. Δηλαδή να καταλήξει η έκθεση να είναι ένα ευχολόγιο χωρίς καμένα ή κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Γιατί εγώ θέλω να έχω μια έκθεση η οποία να είναι ε, συνεπής και ε, προσγειωμένη. Τέλος πάντων θα ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε μάλλον με τους ε, σκιώδεις συγητές ε, για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Κυρία Λίνε, θα, το, θα συζητήσω και μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι οι προτάσεις σας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Τέλος πάντων, πάντως, σας ευχαριστώ όλους. Σε, μία, σε ένα μήνα θα είναι ολοκληρωθεί η έκθεση. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Περές, τον εισηγητή. Θα ψηφίσουμε στις 16 Ιουνίου αφού ακούσουμε τις ε, γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Περιβάλλων ε, Γυναικών κτλ. 2 Ιουλίου ελπίζουμε θα περάσει από την ε, Ολομέλεια. Υπάρχει και ένα σημείο ακόμα στην ημερήσια διάταξη, όπως σας είχα πει, που είναι τα πρακτικά για την εντολή που μας σας δώσατε μέσα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την έκθεση του κυρίου Κασλέρα για την ενεργή γύρανση αν θέλετε στην Ευρώπη και για το έτος ενεργούς γύρανσης το 2012. Δυστυχώς ο εισηγητής δεν μπόρεσε, δεν έχει έρθει ακόμα. Θα είμαι εγώ αναπληρώτρια αλλά πριν σας πω ποια είναι τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης αυτής, να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε τρεις ε, τριμερείς διαλόγους, τρεις τριλόγους τέλος πάντων, ε, σε πολιτικό επίπεδο και δύο τεχνικού χαρακτήρα και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα από την εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας να μας κάνει μία αξιολόγηση από πλευράς του Συμβουλίου όσον αφορά τον τρίλογο αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους από την πλευρά της Προεδρίας του Συμβουλίου ότι εμείς πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Δηλαδή συμφωνήσαμε για το κείμενο της απόφασης αυτής σε πρώτη ανάγνωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερος την Πρόεδρο και τον κύριο Κάσλερ. Με τις προσπάθειές μας, τις κοινέ μας προσπάθειες, μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα και να έχουμε μια καλή μορφή συνεργασίας. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ο καθένας ε, έλαβε υπόψη τις ε, απόψεις των άλλων και έγιναν απαραίτητε παραχωρήσεις. Έχουμε λοιπόν πετύχει το στόχο μας. Και έτσι βλέπουμε ότι θα μπορέσουν στα κράτη-μέλη μέσω της απόφασης αυτής ε, οι υπεύθυνοι και οι φορείς να ξεκινήσουν αμέσως με την υλοποίηση των σχετικών μέτρων. Μάλιστα από το κορεπέρ του, του Μαρτίου ε, πέρασε το πακέτο μέτρων με κάποιες τροποποιήσεις όπως ε, υποβλήθηκαν από την Ουγγρική Προεδρία, στοιχεία που τα παρουσιάσαμε και στις 10 Μαΐου στον τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε ότι στην Ολομέλεια του Ιουλίου θα περάσει χωρίς πρόβλημα το θέμα αυτό και η Ουγγρική Προεδρία στις 17 Ιουνίου θα δημοσιεύσει ενημέρωση. Η Ολομέλεια βεβαίως θα γίνει μετά την ε, Σύνοδο του Συμβουλίου. Αλλά με όλη αυτή τη διαδικασία και εφόσον εγκριθεί και η δική σας απο... η απόφαση και από δική σας πλευράς, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, ελπίζουμε ότι όλε οι συμβαστικέ λύσει θα εγκριθούν ε, και από τη δική σα την πλευρά και σα ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να πω στους συναδελφούς ε, με βάση την εντολή που μας δώσατε η συζήτηση στράφηκε γύρω από τέσσερα σημεία. Πρώτον, ο εισηγητής μας και τον είχατε υποστηρίξει ήθελε να προσθέσει ένα υπότιτλο στο Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης. Ε, an active ε, aging culture. Ε, και να είναι και στα αγγλικά active aging culture. Δηλαδή να έχουμε μια κουλτούρα, μια νοοτροπία ενεργούς γύρανσης. Δεν ήθελα να το βάλει στο τίτλο για να μην είναι υπερβολικά μακροσκελής και χάσει επικοινωνιακά. Ε, το έβαλε στους στόχους όμως και... Αυτό που λέει το θέμα δεν είναι μόνο να επεκταθεί, να παραταθεί ε, ε, ο εργασιακός βίος, αλλά να φροντίσουμε οι ηλικιωμένοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε κοινωνικές υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους ακόμα και εκπαίδευση ε, να μπορούν να έχουν και να μην υπάρχουν διακρίσεις βάρους τους. Ε, το επόμενο φορούσε το πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτού έτους και έγινε ιδιαίτερη μνήα στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των γενεών και στην επιθυμία μας να ενσωματωθούν αυτά, καθώς επίσης και η έννοια της ζωντάνιας, της ζωτικότητας και ε, τους φρίγους για όλους. Άλλο θέμα που μέτρησε πολύ ήταν να δούμε ποιες ήταν οι δραστηριότητες εκείνες που θα μπορούσαμε να φανταστούμε στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γύρανσης και είπαμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι γενναίες, ε, όλοι οι εταίροι, τι εννοούμε, οι κοινωνικοί εταίροι, μικρομεσαίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής και βεβαίως θα ξεχνώ και ε, άλλους πρωταγωνιστές. Και ε, κάτι άλλο που ήταν σημαντικό για τις εκδηλώσεις της χρονιάς αυτής είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και θέματα φύλου αλλά και θέματα προσώπων με αναπηρίες. Περσών και δεν θα μιλήσω ξανά ποτέ για αναπήρους. Είναι άτομα με αναπηρίες. Ε, βέβαια, τίθεται και το θέμα του προϋπολογισμού. Ε, το είχαμε πει και καταφέραμε να κάνουμε το Συμβούλιο να δεσμευτεί και να αναγνωρίσει ότι είναι παράλογο να έχουμε ε, εξαγγείλει ευρωπαϊκό έτος ενεργούς γύρανσης και δεν θέλουμε να βάλουμε καθόλου το χέρι στην τσέπη για να το χρηματοδοτήσουμε. Θα πρέπει και στο προϋπολογισμό κάπου να αντανακλάτε αυτό το κονδύλι για τη χρηματοδότηση της ε, χρονιάς αυτής. Με 5 εκατομμύρια ευρώ που ε, με τον α ή β τρόπο θα πρέπει να αφιερώνονται στις εκδηλώσεις αυτές. Ωραία. Εξαντλήσαμε εδώ λοιπόν την ημέρα. Α, όχι! Ξέχασα. Για να είναι πλήρης η αναφορά αυτή που σας δίνουμε, πρέπει να σας ζητήσουμε να ψηφίσετε για να μπορέσουμε μετά να πάμε στην Ολομέλεια. Όταν θα ολοκληρωθεί το κείμενο, θα είναι το τελικό κείμενο ε, στο Συμβούλιο, θα το έχουν χτενίσει και νομομαθείς, ε, γλωσσολόγοι κτλ. και άλλοι εμπειρογνώμονες. Συμφωνείτε με αυτά που σας προτείνουμε. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά απόχες εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του κυρίου Κάσλερ, τον οποίο εξ ονόματός σας συγχαίρω. Τώρα τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε στις 6 Ιουνίου για μια έκτακτη συνεδρίαση στις 7 η ώρα το βράδυ στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ.